Okay, thank you. Σε ευχαριστώ, Βίτολτ, που προείδρευσε στο προηγούμενο θέμα. Περνάμε τώρα στα σημεία 6 και 7. Μία ώρα έχουμε στη διάθεσή μας για τα δύο αυτά θέματα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και στο όνομα της Ναταλή Λουαζό, που είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής για την Ασφάλεια και την Άμυνα. Θα συζητήσουμε τώρα την ε, ε, ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Κυκλοφόρησε πριν κάποιες εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, και ελπίζω όλοι να είχατε την ευκαιρία να την εξετάσετε. Επικροτώ την ε, δυνατότητα να συζητήσουμε τώρα αυτήν την στρατηγική έκθεση. Σε αντίθεση με την έκθεση του Συμβουλίου για την έκθεση του 2000, ε, σε αντίθεση με την έκθεση του 2019 που ε, υιοθετήθηκε μέσα Οκτωβρίου, αποφάσισα να επικεντρωθώ ε, στη στρατηγική εξέταση των τριών βασικών θεμάτων και να μην κάνουμε απλά μια γεωγραφική περιήγηση. Όπως ε, γνωρίζετε, ε, η πολυμερής προσέγγιση αμφισβητείται και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη για μια πιο ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη. Χρειάζεται να ενεργήσουμε ως γεωπολιτική ε, δύναμη και να έχουμε προορατική προσέγγιση, να δημιουργήσουμε νέες συμμαχίες. Όλα αυτά είναι απαραίτητα και είναι ένα μήνυμα που ακούσαμε και από διάφορους συνομιλητές μας στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη Δευτέρα και Τρίτη. Το δεύτερο είναι ότι για να γίνουμε πιο ισχυροί είμαι επεπισμένος ε, ε, σχετικά με την ανάγκη να ενισχύσουμε ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πυλώνα της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας το Κοινοβούλιο ε, έχει αναπτύξει μια σειρά ε, κατάλληλων εργαλείων και πιστεύω ότι μια τέτοια διάσταση θα είναι ε, θετική για να πετύχουμε το στόχο μας πιο ισχυρής Ευρώπης. Επιπλέον, για να αντισταθούμε σε παγκόσμιες τάσεις είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε την ΚΕΠΑ να ε, έχουμε ε, ενισχυμένη, κανόνα ενισχυ, ε, ενισχυμένης πλειοψηφίας στις ψηφοφορίες και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε υβριδικές απειλές, να εξετάζουμε και τα, τις, τους κινδύνους από την αλλαγή του κλίματος. Ε, τώρα στη Νέα Θητεία αποφασίσαμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό από κοινού με την ΣΕΝΤΕ. Η πρόεδρος Εναταλή Λουαζό ε, θα δώσει το λόγο στον Αρνό Ντανζό ε, για να συζητήσει την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας αμέσως μετά από αυτό το θέμα. Χρειάζεται να επικεντρωθούμε στα μηνύματα κλειδιά, να αποφύγουμε την αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στις δύο ετήσιες εκθέσεις και ε, να μην ε, εισάγουμε εδώ στοιχεία τα οποία εμπίπτουν στην έκθεση για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ε, επικροτώ, μάλλον θα χαρώ πολύ να ακούσω τις απόψεις σας πριν τις τροπολογίες. Θα δώσουμε κατόπιν το λόγο στους ευρωβουλευτές ανάλογα με τις πολιτικές τους ομάδες. Πρώτος ο είναι ο κύριος Πασέσκου από το ΕΛΚ, ε, σωστά το λέω, ή ο Μιχαήλ Γκάλερ. Ο Τράιαν Πασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Κύριε Πρόεδρε, διάβασα την έκθεση, εκτιμώ ιδιαίτερος την προσπάθειά σας ε, να έχετε μια ξεκάθαρη έκθεση για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, λέει ο μιλητής. Έχω μερικές παρατηρήσεις. Ίσως είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να συμπεριλάβουμε στην έκθεση και μια αξιολόγηση. Να αξιολογήσουμε δηλαδή την προστιθέμενη αξία αυτής της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε στο μέλλον να αναπτύξει. Ένα άλλο στοιχείο που φαίνεται απαραίτητο είναι το εξής. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αμυντικών ικανοτήτων του ΝΑΤΟ. Γιατί η έκθεση δίνει την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδιαφέρεται και πολύ για το ΝΑΤΟ. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ως σημαντικό στοιχείο, ως κεντρικό στοιχείο την εταιρική μας σχέση με τον ΝΑΤΟ, ακόμη και τις Ηνωμένε Πολιτείες, αν μου επιτρέπετε. Αυτή η ιδέα, λοιπόν, θα πρέπει να διατρανωθεί στην έκθεση με μεγάλη σαφήνεια. Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας ανάλογα με τις απειλές που αντιμετωπίζουμε όχι να αναπτύξουμε αμυντικές ικανότητες μόνο και μόνο για να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό στρατό. Εντάξει, να έχουμε ευρωπαϊκό στρατό, αλλά θα πρέπει οι αμυντικές ικανότητες να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που απειλούν ε, την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κατά τη γνώμη είναι πολύ σημαντικό. Και τέλος θα σας στείλω κάποιες τροπολογίες Πάντως πιστεύω ότι αυτή η έκθεση που είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη θα πρέπει να είναι τόσο απλή ώστε να την καταλαβαίνουν και τα σχολιόπαιδα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να χρησιμοποιήσουμε πιο απλή γλώσσα για να γίνει κατανοητή και από τους απλούς πολίτες και από τους νέους Ίσως η διατύπωση είναι κάπως συντηρητική. Καλό θα είναι τα έγγραφά μας αυτά να είναι προσιτά σε όλους και ευανάγνωστα. Τι λέτε? Εσείς λέτε ότι η διατύπωση είναι πολύ συντηρητική. Ναι, είπε ότι η, η διατύπωση που χρησιμοποιούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ συντηρητική. Ε, νομίζω ότι είναι εξαιρετική. Δεν βλέπω πολλούς εκτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου που να χρησιμοποιούν την ίδια φρασιολογία. Ναι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ειλικρινά πιστεύω ότι οι εκθέσει μα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστε ώστε να γίνονται αντιληπτέ από όλου, ακόμη και από παιδιά. Ακόμη και αν δεν μα ευχαριστεί μια τέτοια διαπίστωση. Ναι, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει οι συνάδελφοι να αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο της έκθεσης. Πρώτα να ξεκινήσουμε από εμά και μετά να φτάσουμε στους, στον κόσμο. Ναι, αλλά ο κόσμος μας ψηφίζει. Είδατε τι συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν, μας, δεν κατάλαβα τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που καταλήξαμε. Ναι, ναι, αλλά ας δούμε και να καταλάβουμε τι κάνουμε εδώ σήμερα. Οι σοσιαλιστές δημοκρατές δεν ζήτησαν το λόγο, Renew. Τώρα πάμε στον κύριο Μπουτικόφερ και στους πράσινους που θα μιλήσουν πολύ συντηρητικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόθεσή μου ήταν να σας συγχαρώ για το σχέδιο έκθεσης. Όχι λόγω της συντηρητικής ορολογίας που υιοθετεί, αλλά επειδή καταδεικνύει την ποιότητα του να μην είναι κανείς, ε, να μην χρησιμοποιεί τέτοιους περίπλοκους όρους και ε, να μην είναι δύσληπτος. Εγώ προσυπογράφω πλήρως ε, τα όσα μόλις εξηγήσατε σχετικά με την πολυμέρεια. Ταυτόχρονα θυμούμε ότι ο απερχόμενος πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ, μας θύμισε ότι πρέπει να ανακτήσουμε την ικανότητα της τοπικής πολιτικής δραστηριότητας. Και αν το ζητάει από όλους μας, δεν είμαι βέβαιος ότι ως δόκιμη αυτής της ε, ρεαλιστικής πολιτικής προσέγγισης μπορούμε να ηγηθούμε παγκοσμίω. Καλό θα ήταν απλώς να έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε καλοί εταίροι αυτή της ε, πολιτικής προσέγγισης παγκοσμίω και πολυμερός. Πάντοτε δεν εκτίμησα τι τοποθετήσεις της κυρίας Μογκερίνη που ε, ε, περιέγραφε την Ευρωπαϊκή Ένωση ω υπερδύναμη. Αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε αποτέλεσμα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, παρότι βεβαίω αποδέχομαι την απόφασή σας να μην πάμε στο θέμα των παγκοσμίων περιφερειών η στρατηγική διασυνδεσιμότητας δεν είναι ένα περιφερειακό ζήτημα, είναι το πλαίσιο μέσω του οποίου προσπαθούμε να τοποθετήσουμε περιεχόμενο όταν επικαλούμαστε την ε, χρησιμότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής τοποθέτησης. Και έχοντας δει μια θετική ανταπόκριση από τους Ασιάτες εταίρου, ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού Άμπε της Ιαπωνίας. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κρύβουμε την προοδευτική μας συνεισφορά, λέει ο μιλητής. και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής νομίζω ότι πρέπει να πάψουμε να απαιτούμε μονίμως η Ευρώπη να μιλάει με μία φωνή. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί ποτέ αυτό. Εγώ θα ήμουν ικανοποιημένο αν οι περισσότεροι μπορούσαμε απλώς να συνεργαστούμε, να δρούμε από κοινού, αντί μονίμως να προσπαθούμε να πείσουμε αυτούς που έχουν μείνει πίσω και που προσπαθούν να υποσκάψουν την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Να εστιαστούμε δηλαδή σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε μαζί. Ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνουμε άπαντες πάντοτε. Σας ευχαριστώ κύριε Μπιουτικόφερ για τις παρατηρήσεις σας. Από το ID παρακαλώ. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα εκπλαγείτε από τα σχόλιά μου. Διάβασα προσεκτικά αυτήν την ετήσια έκθεση που εγγράφεται σε μια γραμμή σαφέστατη σχετικά με την επικυριαρχία των κρατών και την υποβολή τους ή την υπαγωγή τους στον ύπατο εκπρόσωπο μονίμως περιγράφουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μοναδικό παίκτη εκπρόσωπο σε παγκόσμιο επίπεδο και μιλούμε για την ε, στρατηγική του αυτονομία, για την ε, συνένωση των προσπαθειών των ε, Υπουργών Εξωτερικών σε μια κοινή προσπάθεια σχετικά με τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέγει η εκθεσή σας ρητά ότι το, η διαδικασία λήψη απόφαση πρέπει να κινηθεί από εθνικό σε υπερεθνικό επίπεδο. Σε θέματα ασφάλειας η έκθεσή σας υπογραμμίζει τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και εκτιμάτε ότι η ειδική πλειοψηφία θα μπορούσε να ενισχύσει ε, την δυνατότητα εύκολης λήψης απόφασης ή αποτελεσματικής λήψης απόφασης, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στα δημοκρατικά μας ιδεώδη ε, παρετήτως ούτε τα δικά μας ούτε εκείνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης χαιρετίζεται την απόφαση της Προεδρίας στα πέντε επόμενα χρόνια να δημιουργηθεί μια πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση αμήνης. Είναι αιρετικό, συγχωρήστε μου τον όρο. Τα θέματα της διπλωματίας και της αμήνης σε καμία περίπτωση δεν εμπίπτουν στο ενωσιακό ή το κοινοτικό επίπεδο, αλλά το διακυβερνητικό. Η επικυριαρχία των κρατών μελών στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και αμήνης είναι σαφής. Σας ευχαριστούμε κύριε Ριβιέρ. Εκ μέρους ομάδας Renew, το λόγο έχει Χίλτε Φάουτμανς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά ε, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την εκπόνηση τη σημαντικής αυτής έκθεσης για την εφαρμογή της κοινή εξωτερική Πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Επίσης είναι πολύ επίκαιρη η έκθεση ε, με την έναρξη της εντολής επιτροπή. Επιτροπής. Ε, καλό θα ήταν να ψηφίσουμε την έκθεση πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ο νέος Αντιπρόεδρος Επιτροπής και ε, αρμόδιο για τα ζητήματα εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε ισχυρότερη και πιο ενωμένη Ευρώπη, όπω σωστά λέτε. Θα πρέπει αυτό να είναι το μήνυμά μα και προ τα κράτη-μέλη. Ένα μήνυμα ή τώρα ή ποτέ, αν θέλουμε να είμαστε πιο στρατηγικοί, πιο ε, δυναμικοί και να γίνουμε σημαντικός παράγοντας στο σύγχρονο κόσμο. Γιατί πραγματικά γίνεται μια μετατόπιση του κέντρου δυνάμεων. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μείνουμε στο περιθώριο και σίγουρα αυτό το θέμα ξεπερνάει τα απλά εξωτερικά ζητήματα και την εξωτερική μας πολιτική. Φαντάζομαι θα υποβληθούν αρκετέ κατελές τροπολογίε από τους συναδέλφους. Χαίρομαι πάντως που κάνετε τη διασύνδεση και με τα αμυντικά ζητήματα στην Ευρώπη, γιατί οι εξωτερικέ ε, υποθέσεις, η εξωτερική πολιτική συμβαδίζει με την πολιτική άμυνα. Αυτό που μας λείπει όμως είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε τι ε, μείζονε ε, ε, προκλήσεις, τις δημογραφικές αλλαγές, την αντιτρομοκρατία, τις υβριδικές απειλές, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάποιες παραλήψεις υπάρχουν. Πάντως το Ρινιού θα κάνει το καθήκον του και θα στείλει πολύ εύστοχε τροπολογίε και ευελπιστώ ότι και οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε θα κάνουν το ίδιο. Σα ευχαριστούμε κυρία Φάουτμαν. Η, πλειοψηφία, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια προβλέπεται για τον Ιανουάριο 13 με 16 ε, Ιανουαρίου και ελπίζω μέχρι τότε να έχει αναλάβει και η Νέα Επιτροπή πριν τα μέσα Ιανουαρίου. Ο Τζέφρι Φονόρντερ από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να σας συγχαρώ για την ε, ευστοχία και συντομία σας και το γεγονός ότι κάνετε μια ε, γενική επισκόπηση και όχι περιπτωσιολογική ανάλυση όπως είχαμε στις προηγούμενες εκθέσεις για την ΚΕΠΑ. Και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την παράγραφό σας 17 που εθαρρύνεται την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει προτεραιότητα στην αποτροπή συγκρούσεων, πρόληψη συγκρούσεων, τη διαμεσολάβηση και την ε, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Γιατί εκεί πραγματικά θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια προστιθέμενη αξία. Αυτό που με ενοχλεί και θα σας ε, εκπλήξει είναι η παράγραφη 19, 20 και 21. Εκεί αναφέρεστε στην ειδική πλειοψηφία στα θέματα εξωτερική πολιτική και ασφάλεια και τη σύσταση ενό Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας και μιλάτε και για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Όλε αυτέ οι ιδέε, των παραγράφων 19, 20 και 21 δεν είναι φυσικά καινοφανεί και είναι ε, προσφυλής κάποιων πολιτικών ομάδων, αλλά είναι μηχανισμοί πολιτικής ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διευρύνει το χάσμα με τους διατλαντικούς εταίρους μας, ενώ αντίθετα αυτό που θα πρέπει να τραβήξει την προσοχή μας και να εστιαστούμε είναι η σχέση μας με το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Θα επανέλθω όμως στο θέμα αυτό κατά τη συζήτηση της επόμενης έκθεσης του κυρίου Ντονζόν για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ευχαριστώ, Τζέφρι. Εκ μέρους της Γκουε τώρα δεν έχουμε κανένα ομιλητή. Και περνάμε στο δεύτερο γύρο. Τρεις ε, συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Η Σάντρα Καλνιέτα πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να σας συγχαρώ για την έκθεση. Έχω κάποια σχόλια. Συμφωνώ με τους συναδέλφους εκείνους που αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα της ενίσχυσης και της υπογράμμισης της σημασίας της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, της πιο στενής συνεργασίας με τον ΝΑΤΟ και κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό πόσο ρεαλιστικές είναι οι φιλοδοξίες μας και οι εκτιμήσεις μας της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πραγματικής επιρροής μας στα θέματα των διεθνών σχέσεων. Έχω τα εξής σχόλια. Για μια, η έκκληση για μια πιο αποτελεσματική και στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα τώρα τους τελευταίους μήνες που βλέπουμε πόσο όλο και πιο δύσκολο είναι να έχουμε κοινέ αποφάσεις με τις μετακινήσεις που έχουμε παγκόσμια. Η διεύρυνση, ο Μακρόν, η Ρωσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η εμπορική πόλεμη κτλ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βρούμε μια περίπου κοινή φωνή ως προς αυτά. Άλλη μια ανησυχία για την περιοχή της Βαλτικής τουλάχιστον είναι πώς θα βρούμε έναν πραγματικά δημιουργικό μηχανισμό που θα εξασφαλίσει στα θέματα ασφάλειας και άμυνας την πιο στενή δυνατή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενωμένου Βασιλείου. Χώρα η οποία έχει ισχυρή φωνή και θα πρέπει να βρούμε δημιουργικές λύσεις και για τις διαδικασίες ψήφου χωρίς δικαίωμα βέτο. Και για τα θέματα εξωτερικής ε, δράσης, ε, γειτονίας, ε, ανάπτυξης πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Διότι η γειτονία απαιτεί χρηματική υποστήριξη κατάλληλη. Ευχαριστούμε την κυρία Κανιέτε. Έχω τέσσερις ακόμα ομιλητέ. δεν θα προσθέσω άλλου στον κατάλογο, γιατί περίπου στις και μισή πρέπει να δώσουμε το λόγο στην Άταλη. Δύο λεπτά έκαστο. Ο κύριος Μαγιορίνο, SND, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της έκθεσης αυτής είναι πολύ πιστική έκκληση για μια πιο ισχυρή Ευρώπη και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι μια δραματική επίγουσα αναγκαιότητα. Το να έχουμε μια κοινή προσέγγιση και άποψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφωνώντας προς τα όσα άκουσα από συναδέλφους αυτό το περί μίας κοινής φωνής θα πρέπει να το διατηρήσουμε ως στόχο γιατί η εξωτερική πολιτική, η πολιτική άμυνας, η πολιτική αναπτυξιακή συνεργασίας, μεταναστευτικής πολιτικής πρέπει να είναι καρπός κοινή δουλειά στην Ευρώπη. Και επομένως τα παιδί αυτά πρέπει να είμαστε ακόμα πιο αποφασισμένοι και ακόμα πιο θαραλέοι θα έλεγα. Ακόμα και μιλώντας για τον Ευρωπαϊκό Στρατό, το στρατιωτικό σώμα. η εξασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων που εγώ θα την ε, καθιστούσα ακόμα πιο ρητή ως στόχευση από την ορολογία που έχετε υιοθετήσει στην έκθεση. Επίσης ε, εκφράζω μια ανησυχία σχετικά με τους πόρους. Πρέπει να αποφύγουμε ο στόχος αυτός να οδηγήσει σε ενίσχυση των αμυντικών δαπανών. γιατί εμείς στην ουσία επί τη βάση της χρησιμοποίησης των υφισταμένων πόρων πρέπει να διαρθρώσουμε έναν κοινό αμυντικό στόχο. Και αυτό πρέπει να το βλέπουμε πιστεύω με μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα δεδομένου του γεγονότος ότι πολύ συχνά πόροι που έχουν πιστωθεί για την συνεργασία και την ανάπτυξη που μπορεί να προλαμβάνει την κοινή αμυντική δράση, πολύ συχνά εκτρέπονται προς άλλες στοχεύσεις. Την εξωτερήκευση δηλαδή των συνόρων. Σας ευχαριστώ συνάδελφε, ο Μίχαηλ Κάλερ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ επικροτώ την διάρθρωση της έκθεσης που επιλέξατε. Νομίζω ότι ε, πράγματι αφισβητείται η πολυμερής προσέγγιση και πιστεύω ότι θα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν τον τρόπο που χειρίζονται τα θέματα, ε, το να επιλέγουν να μην έχουμε κοινή δράση για μας. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κατάλληλο μέρος να κάνουμε την έκκληση αυτή. να είμαστε ενωμένοι και εταίροι. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι είμαστε πιο ισχυροί μαζί και ε, να μην ε, δεχόμαστε απλά τις συνέπειες ε, του να μην είμαστε σημαντικός παράγοντας. Επίσης είναι πολύ ε, σωστό που τονίζετε την κοινοβουλευτική διάσταση. Η κοινοβουλευτική διπλωματία συχνά είναι πολύ πιο σαφής ε, στις επαφές που έχουμε με συναδέρφους ή κυβερνήσεις άλλων χωρών και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συμβάλλουμε με λύσεις ε, σε ε, συγκρούσεις που έχουν κολλήσει, όπως για παράδειγμα στα Δυτικά Βαλκάνια. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες αυτές. Επίσης όσον αφορά την ενίσχυση της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, η ειδική πλειοψηφία είναι στόχος, ε, αλλά ε, προσπαθώντας να πετύχουμε τον στόχο αυτό, να θυμόμαστε τις φορές που δεν ε, καταλήξαμε σε απόφαση λόγω ε, τη της μη ύπαρξης ομοφωνίας και νομίζω θα πρέπει να δημοσιεύσουμε ποιοι εμπόδισαν την λήψη απόφασης. Θα υποβάλω πιθανότατα σχετική τροπολογία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μιχαήλ Γκάλερ. Ο κύριος Αλεξάνδρου, παρακαλώ. Благодаря, господин председател. Вземам думата, за Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο για να επιστήσω την προσοχή σας σε μια άποψη την οποία αντιπροσωπεύω εδώ και πολλά χρόνια. Η πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την ε, προσχώρηση νέων μελών στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Για να είμαι πιο ξεκάθαρος, θα πρέπει μια χώρα πρώτα να γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ και μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαράδεκτο να έχουμε μαύρες τρύπες, τις λεγόμενες μαύρες τρύπες ε, στα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ τη Σερβία, για παράδειγμα, είναι χώρες που είναι κατά του ΝΑΤΟ που έχουν ενισχύσει την στρατιωτική τους ε, συνεργασία με την Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν ε, μια εβδομάδα η Σερβία με τη Ρωσία έκαναν ε, στρατιωτικές ασκήσεις ε, χρησιμοποιώντας ε, την τεχνολογία C400 που είναι ε, τεχνολογία που χρησιμοποιούν η Σερβία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία. Πρόκειται για πυράβλους που που μπορούν να χτυπήσουν τις χώρες αυτές. Και διπλωμάτες είχαν επαφές με τις μυστικές μας υπηρεσίες. Πριν λίγες μέρες ο Βλάντιμιρ Πούτιν ε, έδωσε βραβείο, ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία της χώρας σε έναν Βούλγαρο που ανοιχτά υποστηρίζει μια ε, οργάνωση που είναι κατά του ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τονίσουμε το ρόλο της ε, Ρωσίας ε, ως ε, χώρα αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Επίσης, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει πρώτα να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Τέλος. Ευταίως ο κύριος Σικόρσκι. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε, πολύ χρήσιμη έκθεσή σας και σε αυτούς που θέλουν μια λιγότερο ενωμένη Ευρώπη με μεγαλύτερη επιρροή, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό είναι αντιφατικό. Δεν γίνεται στο σύγχρονο κόσμο. Αν θέλουμε μια Ευρώπη με περισσότερη επιρροή, θα πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι και να δρούμε από κοινού. Και μου άρεσαν οι ιδέες σας και για την ειδική πλειοψηφία και η ιδέα του Μάικλ να κατονομάσουμε χώρες που παραβιάζουν την ομοφωνία που αποκλίνουν. Ε, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κοινή πολιτική ακόμη και όταν ε, καταλήγουμε σε συνένεση, σε ομοφωνία. Γιατί συμφωνούμε σε κάτι στο Συμβούλιο και κατόπιν τα κράτη-μέλη κάνουν του κεφαλιού τους ε, επιτρέπουν τάχα στον στην είπατε εκπρόσωπο να ακολουθήσει μια πολιτική, αλλά έχουν και τις δικές τους ιδέες κατά μέρους, είτε για την Ουκρανία, τη Ρωσία, ε, το Ιράν, ε, τη σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ακόμη και όταν έχουμε καταλήξει σε κοινή θέση και έχουμε συμφωνήσει, παρόλα αυτά δεν δρούμε ενία Θα ήθελα λοιπόν ε, να είμαστε κάπως πιο κατηγορηματικοί στην έκθεση και να πούμε ότι τα κράτη-μέλη καταστρατηγούν τις συνθήκες. Γιατί Έχουμε δεσμευτεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας και έχουμε ε, δεσμευτεί να δρούμε από κοινού. Οπότε θα πρέπει να αφήνουμε κατά μέρο ε, ε, τα εθνικά συμφέροντα. Γιατί ο χώρο προάσπιση των εθνικών συμφερόντων είναι το Συμβούλιο. Από τη στιγμή όμω που το Συμβούλιο έχει καταλήξει σε κοινή θέση, θα πρέπει να στηρίζει πιστά και αφοσιωμένα την είπατε για την άσκηση αυτή τη πολιτική. Και ε, βέβαια, μετά χρησιμοποιούνται οι εθνικοί υπουργοί για να, γίνουν, ε, να ασκηθούν πολιτικές ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η πρακτική της Lady Άστον όταν ήταν ύπατη εκπρόσωπος. Και ελπίζω και ε, η ο διάδοχος μάλλον της κυρίας Μογκερίνη να επιστρέψει σε αυτή την πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και τις χρήσιμες παρατηρήσεις. Ε, την Παρασκευή σε 11 το πρωί λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες. Στις 18 Νοεμβρίου θα τις εξετάσουμε. Η συνεδρίαση με τους και ηγητές θα γίνει ε, στην 47η-8η ε, εβδομάδα. 4 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και αν όλα βγουν κατευχήν στις 13 με 16 Ιανουαρίου στην Ολομέλεια του Στρασβούργου θα ψηφίσουμε και την έκθεση. Και θα δώσω το λόγο τώρα και την Προεδρία μάλλον στην Αταλή Λουαζό για να προεδρεύσει στο σημείο 7. Θα μιλήσω γαλλικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσουμε τώρα για την ετήσια έκθεση της υλοποίησης της ε, κοινή ε, πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας. Πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Ντάνζο. Ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα. Η υποβολή των τροπολογιών για την έκθεση πρέπει να γίνει πριν από την Παρασκευή αυτή, 8 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Θα εξετάσουμε στην ΑΦΕΤ 18 Νοεμβρίου τις τροπολογίες με ψήφο στην ΑΦΕΤ 4 ε, Δεκεμβρίου και εκτάκτος έχουμε ένα χρονικό παράθυρο στην ΑΦΕΤ ώστε να μπορέσουμε να πάμε στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο του 20. Ο αγνό των Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Μιλούμε για μια ετήσια έκθεση για την υλοποίηση, την εφαρμογή της κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Δηλαδή το πλαίσιο είναι ήδη περιορισμένο και το λέω αυτό διότι υπάρχει μια τάση μεταξύ κάποιων συναδέλφων για αυτά τα θέματα να έχουμε ευρύτατες γεωπολιτικές αναλύσεις και παρατηρήσεις για το σύνολο του κόσμου και των κρίσεων. Δεν είναι ο στόχος έκθεσης αυτής. Μιλούμε για την εφαρμογή των στοιχείων που εντάσσονται στη συνθήκη για την κοινή αυτή πολιτική. Δηλαδή το εύρος της έχει περιοριστεί εγώ δεν έχω καμία διαφωνία να έχουμε ευρύτατες συζητήσει. έχουμε πολλές δηλαδή, αλλά δεν είναι η δουλειά μας σχετικά με αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη έκθεση. Τώρα, να σας ε, μιλήσω για την έκθεση αυτή της εφαρμογής της πολιτικής αυτής που είναι μια πολιτική μετριοπαθής, περιορισμένου πεδίου, γιατί παραμένει εδώ το θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών διακυβερνητικής δηλαδή προσέγγισης, εμείς δεν προσπαθούμε να μεταβάλουμε κάτι τέτοιο, αλλά να αξιοποιήσουμε τα κοινά εργαλεία που έχουμε στη θέση μας. Και τα οποία είναι αποστολές και επιχειρήσεις, 16 έχουμε αυτή τη στιγμή, πολιτικές και στρατιωτικές, και προσπαθώ να επιφέρω μια, απο, μια πλήρη αξιολόγηση για κάθε μία από αυτές τις αποστολές, οι οποίες ε, με πολύ επαγγελματικό τρόπο ε, διεξάγονται και από στρατιωτικό προσωπικό και από πολιτικό προσωπικό. Ο αντίκτυπος όμως των προσπαθειών αυτών είναι τελείως άνισος. Και μπορούμε να έχουμε εδώ ουσιαστική βελτίωση. Ιδιαίτερα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των αποστολών και των επιχειρήσεων αυτών για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά του. Αυτό το λέμε εδώ και καιρό. Είναι δύσκολο να το πετύχουμε στην πράξη, αλλά είναι μια διεκδίκηση που πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε. Προσπάθεια. Για την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκή Ένωσης γνωρίζω ότι είναι θέμα προκαλεί συζητήσει. Και επανέρχομαι συχνά στο κείμενο σε αυτό διότι πρόκειται για μια έννοια που σήμερα βλέπουμε στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι σχετικά με αυτό, δεν είναι προφανές για όλους. Οι έννοιες αυτές δεν είναι προφανείς και ίσως πρέπει να γίνονται πιο συγκεκριμένες και είναι το αποτέλεσμα δύο συμπερασμάτων ή της σύγκλησης δύο συμπερασμάτων. Καταρχάς, η τη συγκληση δυο συμπερασματων καταρχας η υποχωρηση του στρατηγικού μας περιβάλλοντος η οποία οδηγεί τους Ευρωπαίους σε μια αναπροσαρμογή της στρατηγικής τους σκέψης. Δεν μπορούμε πλέον, όπως είχαμε κάνει επί δεκαετίες, να εξαρτόμεθα από την, το διμερές σύστημα και από συμμαχίες που έχουν πλέον αποδιαρθρωθεί, αποδομηθεί. Ε, είμαστε αντιμέτωποι με κρίσεις γύρω-γύρω και τα μέσα μέσω των οποίων διαχειριζόμασταν τα θέματα ασφαλείας 60 χρόνια τώρα είναι πλέον υπό απειλή. Δεν λέω ότι έχουν εξαφανιστεί, δεν λέω ότι είναι ασήμαντα, αλλά βλέπουμε ξεκάθαρους περιορισμούς. Οι ίδιες συμμαχίες αμφισβητούνται από το εσωτερικό, όταν οι πιο σημαντικοί μας σύμμαχοι, οι Ηνωμένε Πολιτείε, προχωρούν στην πολιτική που προχωρούν με τρόπο τόσο απότομο και ε, ευνηδιαστικό όταν στη συμμαχία έχουμε τον κύριο Ερντογάν τότε κανείς μπορεί να αμφισβητεί το κατά πόσον είναι συμμαχία αξιών το ΝΑΤΟ όταν έχουμε ως σύμμαχο τον κύριο Ερντογάν. Επομένως υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, μία αμφιβολία που πρέπει να οδηγήσει τους Ευρωπαίους ως κράτη αλλά και συλλογικά στη μεγαλύτερη αυτονομία στην μικρότερη εξάρτηση από άλλους, όποια και να είναι. Γιατί δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις σε ζώνες που δεν δηλώνονται ως προτεραιότητα από τους συμμάχους μας. Δηλαδή στα, στο νότο όπου έχουμε ιδιαίτερη αστάθεια, έχουμε εταίρους, έχουμε συμμάχους που δεν έχουν προτεραιότητα να δουν, να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις και την αστάθεια σε αυτά τα εδάφη. Δεν μιλώ για απόλυτη και πλήρη ανεξαρτησία, γιατί αυτό δεν θα ήταν καθόλου ρεαλιστικό, μέσω πρόθεσμα τουλάχιστον, αλλά μια αυτόνομη τουλάχιστον ικανότητα αξιολόγησης, ανάλυσης των καταστάσεων και δυνατότητας παρέμβασης αυτόνομης. Και αυτό είναι φιλόδοξο. Είναι κάτι που δεν έχουμε σήμερα σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά είναι μια φιλοδοξία με την οποία πρέπει να οπλιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν λέω Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ τα κράτη-μέλη. Τα κράτη που θα πρέπει να καταβάλουν την προσπάθεια. Χρησιμοποιώντα κάποια μέσα που έχουμε στη θέση μα ενωσιακά. Σε γενικέ γραμμέ, αυτέ είναι οι θεματικέ τη έκθεση. Επανέρχομαι στα καινούργια μέσα που έχουμε το 2016. Μερικά από αυτά ήταν συνθήκη, όπω η ε, δομημένη μόνιμη συνεργασία. Έχουμε σημειώσει πρόοδο εκεί σημαντική θα έλεγα ότι και θεωρητικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα γιατί φαίνεται να είμαστε πλέον έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα ταμπού του παρελθόντος ότι δηλαδή η Επιτροπή δεν μπορεί να χορηγεί κονδύλια στα θέματα μήνης και όταν συζητούμε για το ταμείο της μόνιμης αυτής συνεργασίας που κανείς δεν ήθελε να τον ενεργοποιήσει πλέον μπορούμε να συζητούμε την ενεργοποίησή του. Τώρα το ύφο έκθεσή μου θα το επικρίνουν κάποιοι σίγουρα και είμαι σίγουρο ότι θα εμπλουτιστεί η έκθεση από διάφορε τροπολογίε και παρατηρήσει και προσθήκες δικέ σα. αλλά η διαρθρωμένη μόνιμη συνεργασία 47 έργα σε 27 χώρε. Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορούμε να μιλούμε για μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία για να μπορούμε να προχωρήσουμε με, με κράτη εθελοντές. και το Ταμείο Αμήνης είναι προς το παρόν θεωρητικό. Έχουμε προβλέψεις ε, κονδυλίων, πορών, έχουμε δεσμεύσεις, αλλά δεν είμαστε σε καμία περίπτωση σε μια επιχειρησιακή ετοιμότητα ε, για το ταμείο αυτό και ο διάβολος πάντοτε κρύβεται στις λεπτομέρειες. Όπως γνωρίζετε, η εφαρμογή είναι πλέον, ε, είναι ακόμα μάλλον η πρόθεση και όχι η πραγματικότητα. Κάποιοι ίσως ε, επίση να επικρίνουν και με αυτό θα κλείσω ε, τις ε, πολύ λίγες μνήες στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το κοινοβούλιο μας, τα κοινοβούλια μας πρέπει να διαματίσουν το ρόλο τους. Και δεν πρέπει να αναρωτιούνται πλέον για την αρμοδιότητά τους στο αμυντικό πεδίο. Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τις αποφάσεις, είναι σαφές, αλλά δεν έχουμε εδώ υπό τη συνθήκη τα νομικά εργαλεία που χρειαζόμαστε για να λαμβάνουμε αποφάσεις οι οποίες παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εγώ θέλω πάντοτε να είμαι ρεαλιστής στις προσεγγίσεις μου αυτές. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι σίγουρα ε, αποτελεσματικά εξασκούμε τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα αντί να διεκδικούμε ή να ζητούμε άλλες προκειμένου να διενεργούμε μια σωστή κοινοβουλευτική επιτήρηση ή παρακολούθηση των μέσων αυτών της πολιτικής αυτής. Δηλαδή του ελέγχου των αποστολών της συνεργασίας που υλοποιείται εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εκεί έχουμε ρόλο και πρέπει να είμαστε πιο δραστήριοι και πιο αναγνωρισμένοι. αντιεθνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν προσωπικό εθνικό και εκεί σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεκδικήσει το ρόλο του εκεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντανζό. Θα δώσω τώρα το λόγο σε ένα πρώτο γύρο συζήτησης στους κοιόδης ηγητές. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Αρακόβατς, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Είναι εδώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα ως και ο να συγχαρώ τον κύριο Ντανζόν για την πολύ άρτια του έκθεση. Ε, είναι πολύ διεξοδική και τεκμηριωμένη. Απ' την άλλη λυπάμαι που το Συμβούλιο δεν ε, τήρησε το καθήκον του και δεν έστειλε έγκαιρα την ετήσια έκθεση του για την ΚΕΠΑ. Συμφωνώ ότι η ΚΕΠΑ, λέει ο μιλητή, η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, ε, θα συμβάλλει στη μεγαλύτερη ολοκλήρωση, ενθαρρύνοντα την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στο παγκόσμιο προσκήνιο και να γίνει σημαντικό παράγοντα. Γι' αυτό θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να περάσει τα θέματα ΚΕΠΑ από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία γιατί κάτι τέτοιο το προβλέπει και το επιτρέπει η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μακροπρόθεσμα είμαι υπέρ της ιδέας της σύστασης ενός ευρωπαϊκού στρατού. Παρόλο που γνωρίζω ότι υπάρχουν ακόμη και στην αίθουσα αυτή πολέμοι της πρότασης και καταδικάζουμε την στρατιωτική επέμβαση της και τη της Ρωσίας στην Κρυμαία, στη χερσόνησο της Κρυμαίας και στηρίζουμε την ε, εδαφική ακαιρεότητα, ανεξαρτησία και κυριαρχία της Ουκρανίας. Και στοχευμένα περιοριστικά μέτρα μπορεί να είναι αποτελεσματικά, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν θα πρέπει να επηρεάζουν αθώους ή να τους πλήττουν και θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ΚΕΠΑ. Και επίσης ε, να έχουμε πολυμερείς ε, διαπραγματεύσεις για, τη, για τα πυρηνικά και να ε, αντιμετωπίσουμε υβριδικές απειλές όπως είναι οι προπαγανδιστικές εξαιρετικές παραπληροφόρησης. Επίσης, να στηρίξουμε τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΕΠΑ και να εξάρουμε τα επιτεύγματα τις τελευταίες ε, με την ενίσχυση της ΚΕΠΑ και ελπίζω η πρόοδος να συνεχιστεί και στο μέλλον. Αποουσιάζει ο κύριος Πάετος και ο δισηγητής της ομάδας Ρινιού. Ε, για τους πράσινους η κυρία Νόημαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Ντονζόν για την πολύ πλήρη ε, και ευρία έκθεσή σας για την ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Υπάρχει μια σειρά θεμάτων στα οποία ε, συμφωνούμε μαζί σας, ε, όπως ε, αυτά που αφορούν τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων καθώς και την προσέγγιση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να έχουμε μια πιο ικανή, μια πιο αποτελεσματική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ε, δεν θα σας εκπλήξει όμως ότι έχουμε και μια σειρά τροπολογιών ε, στην έκθεσή σας ε, και θα σας αναφέρω τα θέματα ε, ε, που θα πραγματεύονται. Αναφερθήκατε στη στρατηγική αυτονομία. Ε, εμείς δεν είμαστε βέβαιοι αν θα πρέπει να είναι στόχος ή απλά, αν θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός ή απλά να είναι ένα μέσο για την κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η αποτελεσματική, η υπεύθυνη κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ε, που να βασίζεται σε αξίες για να είναι σημαντικός και αξιόπιστος εταίρος η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο, στη διεθνή σκηνή. Έχετε δίκιο ότι το να μπορούμε να ενεργούμε αυτόνομα ε, μπορεί να αποτελέσει τρόπο να πετύχουμε το στόχο αυτό, αλλά η δημιουργία συμμαχιών, η συνεργασία και η ενίσχυση της πολυμερούς προσέγγισης θα πρέπει επίσης να είναι τρόποι να πετύχουμε το στόχο αυτό. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι ότι το 90% ε, του κειμένου σας επικεντρώνεται στην ε, βιομηχανία άμυνας σε αμυντικές ε, δομές. Ωστόσο, νομίζω ότι ο πυρήνα τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την πολιτική πλευρά της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις 11 ε, πολιτικές αποστελές μας, ε, διότι όταν ενεργούμε υπό την αιγίδα της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας πρόκειται κυρίως για πολιτικές και όχι στρατιωτικές αποστολές. Τρίτη παρατήρηση. τι αποτέλεσμα πετυχαίνουμε με τις αποστολές αυτές ε, και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο σε τι βαθμό ε, μπορούμε να ε, εξετάσουμε με τρόπο διαφανή το τι κάνουν εκεί οι αποστολές μας. Νομίζω ότι ο καθένα που συμμετέχει στι αποστολέ αυτέ θέλει να βελτιώσει την κατάσταση στι χώρε αυτέ. Πολλοί διακινδυνεύουν τη ζωή του για να το πετύχουν αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίζετε αυτό. Ωστόσο, εάν δούμε το αποτέλεσμα ε, των αποστολών αυτών ε, και τις ε, ενέργειες που αναλαμβάνουν, μερικές φορές βλέπουμε ότι συνεργάζονται με παράγοντες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και που έχουν παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Και δεν το λέω αυτό ω επιχείρημα κατά των αποστολών αυτών. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικές. Είναι πολύ σημαντικό όμως εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο και αλλού να ε, εξετάζουμε πιο προσεκτικά τι, κάνουμε και να, τι κάνουν και να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια των αποστολών αυτών. Ε, για παράδειγμα, στο ε, Ιράκ θα πρέπει να εξετάσουμε τι κάνει στην παρούσα κατάσταση. Μία τελευταία παρατήρηση πριν τελειώσω. Αναφερθήκατε στην πιο στενή συνεργασία, στην έρευνα και ανάπτυξη των ε, αμυντικών δυνατοτήτων. Ε, θέλουμε να φροντίσουμε να έχουμε τον ίδιο βαθμό συνεργασίας και εποπτείας κατά την εξαγωγή των όπλων, ιδιαίτερα όσων ε, χρηματοδοτούνται από μηχανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές λοιπόν είναι αυτά είναι τέσσερα θέματα πάνω στα οποία θα υποβάλουμε τροπολογίες και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μία ολοκληρωμένη εκθέση που θα συμβάλλει στην ενίσχυση τη κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να είστε πιο συνοπτικοί και λακωνικοί στι ομιλίε σα. Από σεβασμό προ του ε, επόμενου ομιλητέ, γιατί και αυτοί δικαιούνται λίγο χρόνο. Άλλωστε, μέχρι την Παρασκευή έχετε χρόνο να καταθέσετε τροπολογίε στο σχέδιο έκθεση. Εκ μέρου τη ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία, το λόγο κύριο Ριβιέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Αρνόντα Ανζόν για το έργο του. Ε, εκτιμώ ιδιαίτερα στα εισαγωγικά του σχόλια, ε, όπου υπενθύμησε τον περιορισμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά και είπε ότι θα πρέπει να τηρήσουμε πιστά τις συνθήκες. Και όμως η έκθεση δείχνει ότι είναι καρπό συνένεση, συμβασμού, γιατί παρόλα αυτά εντάσσεται στην θέληση δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής που θα αντικαταστήσει με το πρόθεσμα της ε, αμυντικής πολιτικής των κρατών μελών και μιλάει για μια ολοκλήρωση των αμυντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια μιλάει για ε, στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάτε ε, για την μια απομάκρυση από τον, από τον ΝΑΤΟ, ενώ ε, κανονικά θα πρέπει να είναι αυτή η έπεση στην εταιρική μα σχέση. Δεν θα πρέπει να είμαστε ουραγοί, λέτε, ε, ως προς τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε, ενώ οι αμυντικές μας δαπάνε είναι πολύ μικρότερες. Επίσης, η συνθήκη τη Λισαβόνα θέλει να τροποποιήσει τους μηχανισμούς ε, ε, και μάλιστα θέλουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά της, λέμε, τα τελευταία χρόνια. Ε, σε σχέση με την έκθεση Μακάλιστερ, η δική σας έκθεση ουσιαστικά ξεπερνά τις ευρωπαϊκές συνθήκες και βάζετε τη διπλωματία και την ε, άμυνα στο περίμετρο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα θέλετε να την υποτάξετε στον κανόνα της ειδικής πλειοψηφία και όχι στην ομοφωνία που ισχύει τώρα. Ε, κάνετε έναν απολογισμό και των αποστολών σε ό,τι αφορά την ε, ε ναυτική επιχείρηση, θαλάσσια επιχείρηση Σοφία, Euronav Met, δεν μιλάτε όμως ότι στόχος της είναι η συστηματική απόθεση και επαναπατρισμός των μεταναστών στην προέλευση, στη χώρα προέλευσή τους ή στη χώρα από την οποία ξεκίνησαν. Επίσης, ε, μιλάτε για την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της Ευρωπαϊκής Άμυνας, δηλαδή την ε, απειλή ουσιαστικά των ε, ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών. Αυτό όμως μας απομακρύνει από την αρχική μας προσέγγιση της διακρατικής συνεργασίας για τα αμυντικά θέματα. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα, εκφράζεται την ευαρέσκειά της για τα 13 δισεκατομμύρια που έχουν προγραμματιστεί. Αυτό όμως είναι μια πρωτοβουλία για μια κοινοτικοποίηση του αμυντικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα τίθεται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα καταθέσουμε φυσικά πολλές τροπολογίες προκειμένου τα αμυντικά ζητήματα να παραμείνουν όχι στο κοινοτικό πεδίο αρμοδιοτήτων, αλλά να παραμείνουν στο διακυβερνητικό πεδίο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανόρντεν για το ECR, παρακαλώ, λέει η πρόεδρος. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Πρόκειται για μια προσεκτικά διατυπωμένη έκθεση. Ε, δεν θα περίμενα τίποτα λιγότερο από τον κύριο Ντανζόν. Όχι ότι αναγκαστικό σύμφωνο βεβαίως με, τις, ε, με όλες τις προσεγγίσεις τους μιλούμε για στρατηγική αυτονομία. Ε, είναι σαν να λέμε ότι η ασφάλεια και η άμυνα θα έπρεπε να είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ διαφωνώ. Και ότι αν είναι να επιτύχει τις κρατικές φιλοδοξίες της πρέπει να έχει στερεωτικά μέσα. Αυτό έχει μια λογική από μόνο του, αλλά εγώ διαφωνώ προς τη στόχευση. Νομίζω ότι σκοπίμως επιχειρείται εδώ μια ακόμα μεγαλύτερη απόκληση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών που δεν μπορεί παρά να ικανοποιεί τους αντιπάλους μας, τους εχθρούς μας, λέει ο μιλητής, και μπορούμε να επικαλούμαστε τη στρατηγική αυτονομία όσο τα πράγματα δεν είναι υπερβολικά δύσκολα. Γιατί όταν είναι δύσκολα τα πράγματα, όταν γίνονται δύσκολα, τότε καλούμε τους συμμάχους μας, τους Αμερικανούς, να τα λύσουν και δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σημαντική κλίμακα χωρίς τη συμμετοχή των Αμερικανών. Δηλαδή φαντάζομαι κάποιε αποστολές ίσως περιορισμένες αντιτρομοκρατική ε, προσπάθεια, αλλά σίγουρα όχι πολεμικές επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε και στην παρατήρηση της έκθεσης του κυρίου Μακάλιστα για προληπτικές δράσεις, για ανθρωπιστική δράση και επιχειρήσεις, όπου εκεί πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι χρήσιμη και συμπληρωματική προς τον ΝΑΤΟ. Δεν θα έπρεπε να προσπαθούμε εδώ να δημιουργήσουμε αμυντικές δομές ε, που όχι να, να ανταγωνίζονται αλλά να απειλούν διαιρέσει εντός του ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ. Ε, για την ΚΟΕ παρακαλώ, μη Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμένα με απογοητεύει η έκθεση αυτή και θα το εκφράσω μέσω τροπολογιών. Μου φαίνεται ένα σύγχρονο μανιφέστο απεικιοκρατίας για μόνιμο πόλεμο, χωρίς ε, κανένα σεβασμό στο 2-4 άρθρο τρομένων εθνών, ε, σχετικά με την επικυριαρχία των αναξαρτήτων χωρών. Ε, καλούμε διάφορες χώρες να προστατεύσουν τα ούτως αποκαλούμενα συμφέροντά μας, διαφορώντας για τους πόρους τους και με τρόπους που θα μπορούσαν να εκφραστούν ως ρατσιστικοί και εκφράζοντας τους μετανάστες ως απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς ούτε και μία φορά να αναγνωρίζουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αποσταθεροποίηση πολλών χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Εμείς δεν τα κάναμε όλα αυτά στη Λιβύη, στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, δεν στείλαμε εκατομμύρια ευρώ αξίας ε, πολεμικό υλικό σε διάφορους ε, αιμοσταγείς δικτάτορες. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν στοιχεία, θα χρειαζόμασταν λίγο περισσότερο κοινό νου αντί να προσπαθούμε να έχουμε ε, συμμετοχή σε μια μεγαλύτερη συμμαχία με πιο σύγχρονα και δολοφονικά όπλα και με μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν υψηλότατη κερδοφορία πουλώντας ε, δολοφονικά όπλα σε δικτάτορες και στην εξόριξη πόρων που θα έπρεπε να μένουν στο χώμα, στον πλανήτη και προκαλώντας δυστυχία στους λαούς, ε, στον κόσμο και συνεργασίες που δεν σέβονται καμία ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις οποίες φιλοδοξούμε να ολοκληρώσουμε. Η προτεραιότητά μας θα έπρεπε να είναι η αποτροπή των κρίσεων και όχι η ενίσχυση προς την αμυντική βιομηχανία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έχω πολλούς ομιλητές που ζητούν το λόγο. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας ικανοποιήσω όλους. γιατί έχουμε και το επόμενο θέμα στη διάταξη και θα έπρεπε να έχουμε ήδη ξεκινήσει με αυτό. Επομένω λίγα λεπτά ακόμα για τέσσερις ομιλητέ θα έχουμε. Παρακαλώ τους τέσσερις αυτούς ομιλητέ να μείνουν στο ένα λεπτό και τις ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ο κύριο Γκάλα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Ανώ για την ε, πολύ καλή έκθεση του. Σημερίζομαι την ισορροπημένη προσέγγιση του όσον αφορά τις πολιτικές αποστολές και τα στρατιωτικά μέσα. Επίσης όσον αφορά τη στρατηγική αυτονομία μας και τις αποτελεσματικές αποστολές. Τους επόμενους μήνες περιμένουμε επιτέλους να ε, ορίσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τη στρατηγική αυτονομία. Ε, και να έχουμε πολιτική δήλωση σχετικά με την κινητική πολιτική ασφάλειας ε, και άμυνας και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Επίσης, ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ε, επικεντρωθούμε και στην ε, βιομηχανία άμυνας και όσον αφορά τις ε, τρίτες χώρες θα πρέπει να επιβάλλουμε προϋποθέσεις και αποκινούμε τις Ηνωμένε Πολιτείες να πετύχουμε την αμοιβαιότητα όσον αφορά τα προϊόντα της βιομηχανίας άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αμερικανική αγορά. Επίσης ε, έχουμε ε, μεγάλη διατλαντική εξάρτηση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή και ε, αμερικανική βιομηχανία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε ρεαλιστικά την βιομηχανία όπλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσουμε άνοιγμα της Αμερικανικής αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σούστερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βρίσκω και εγώ ενδιαφέρουσα την έκθεση και ε, συμφωνώ το ότι χτίζεται σε μια στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο θα πρέπει να έχουμε ορισμό του όρου αυτού. Είναι πολύ ανοιχτή η έκθεση, δεν ε, αναφέρει πιο συγκεκριμένα πώς ε, θα διαμορφωθεί η σχέση μας ε, με το ΝΑΤΟ ή τον ε, ΟΗΕ. Έχουμε στρατιωτικές παρεμβάσεις μόνο μετά από εντολή του ΟΗΕ ή μιλάμε για τελείως ανεξάρτητη στρατηγική δυνατότητα και ποια είναι η σχέση ανάμεσα στους μηχανισμούς επίλυσης κρίσεων, τους στρατιωτικούς και τους πολιτικούς. Και γιατί χρειαζόμαστε όλο και, περισσότερους, ε, όλο και περισσότερο εξοπλισμό. Ε, μήπως ε, έχουμε σπατάλη δισεκατομμυρίων που θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε με πολύ καλύτερο τρόπο. Αυτά παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καλνιέτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα αναφερθώ κυρίως θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως σε αυτή την πρωτοφανή αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Από τα 590 εκατομμύρια περνάμε στα 13 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 22 φορές αύξηση. Πάνω από 20 πλάσια αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο δημοσιονομικό επταετή κύκλο. Αυτό που με προβληματίζει είναι έχουμε την ικανότητα να απορροφήσουμε τόσο εκθετική αύξηση του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια πολύ αποτελεσματικά για την έρευνα και την άμυνα. Και για όλες τις νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, που, σχε... σχετίζονται και με πολύ μεγάλη αύξηση των δαπανών, για όλες αυτές τις αποστολές θα πρέπει να θεσπίσουμε ξεκάθαρους όρους ε, και κριτήρια που δεν υπάρχουν πάντα. Για παράδειγμα, θέλουμε μια αποτελεσματική διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού, συμμετοχή των κρατών μελών, αντίκτυπο στις πραγματικές ε, ανάγκες ε, ικανότητων και επίση λογοδοσία του Συμβουλίου, η πλαίσιο λογοδοσία για το Συμβούλιο. Όλα αυτά είναι σημαντικέ προποθέσει. Και ο τελευταίο ομιλητή στο γύρο αυτό, κύριο Γκέτα. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ ε, και εκ μέρους της ε, ομάδας μου, του Renew Europe. Να προσθέσω λοιπόν και τα δικά μας συγχαρητήρια και επένους προς τον ε, συντάκτη της έκθεσης, τον κύριο Ντανζόν. Επίσης, θα ήθελα να θυμηθούμε όλοι εδώ ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπανούν από κοινού σε στρατιωτικά θέματα ε, σε κονδύλια από τη Ρωσία για αποτελέσματα όμως που είναι πραγματικά απογοητευτικά, αξιοθρύνητα. Και αυτή η απλούστατη σύγκριση μεταξύ ημών και των Ρώσων θα πρέπει να μας ε, εμψυχώσει και να μας παροτρύνει να καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες συντονισμού των ενεργειών μας και των προσπαθειών μας. Όταν κάποιοι συνάδελφοι μας λένε ότι δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε σήμερα χωρίς το ΝΑΤΟ, βεβαίως αγαπητοί συνάδελφοι, ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς ε, ε κάνουμε τη συζήτηση και εκεί έγκυται ε, το δράμα μας. Γιατί με τον παρόντα πρόεδρο ε, των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά γενικώ με τις Ηνωμένες Πολιτείες ασχέτως πρόεδρου, εδώ και χρόνια αμφισβητούν τη διάρκεια και την ε, ε, ευρωστία της ε, Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Οπότε, αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς το ΝΑΤΟ και αν δεν έχουμε κοινή αμυντική πολιτική, δεν θα έχουμε ουσιαστικά στο μέλλον καμία άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, συμμερίζομαι το σχόλιο του Ντανζόν για τα όρια της προσπάθειάς μας και το πλαίσιο που μας δεσμεύει. Αλλά δεν κατάλαβα αυτό που μας είπε πριν από λίγο προφορικά και δεν αναφέρει στην έκθεση. Ελπίζω να μην κατάλαβα καλά και να τον παρεξήγησε. Είπε ότι δεν θα έπρεπε να εκφράζουμε επιθυμίες ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μην εκφράζουμε τις επιθυμίες μας για την εξέλιξη της ε, αμυντικής πολιτικής, γιατί δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Ναι, όντως, ισχύει. Δεν έχουμε τις δημοσιονομικές εξουσίες ε, και από αυτή την άποψη δεν έχουμε την ε, σχετική αρμοδιότητα. Αλλά γιατί να μην ε, εκφράζουμε τις επιθυμίες μας και να μην κάνουμε προτάσεις. Έχουμε απόλυτο δίκιο και να μην έχουμε καθήκον να εκφράζουμε τις επιθυμίες μας και να υποβάλουμε προτάσεις. Σας ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο για πολύ σύντομο όμως διάστημα στον κύριο Ντανζό. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα γιατί ε, μπορούν οι συνάδελφοι με τις τροπολογίες τους ε, που θα συζητήσουμε στις 18 Νοεμβρίου να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμβάλλουν στην έκθεση. Ε, φυσικά δεν με εξέπληξαν οι θέσει των διαφορών ομάδων. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία. Ως προς το τελευταίο σχόλιο του κύριου Γκέτα. Δεν με παρεξήγησατε. Με καταλάβατε πολύ καλά. Μια χαρά. Φυσικά είμαστε εδώ και για να εκφράζουμε επιθυμίες και φιλοδοξίες και για να υποβάλουμε προτάσεις. Απλώς Είπα ότι πολύ συχνά, και δεν αναφέρομαι σε εσά γιατί είστε νέο εκλεγή βουλευτής, πολύ συχνά τέτοιε συζητήσει ε, ήταν ευκαιρία και ε, δυνατότητα να υποβληθούν προτάσεις που ναι μεν ήταν θεωρητικά ενδιαφέρουσες αλλά τόσο άσχετες με τις πραγματικές μας αρμοδιότητες που ήταν ουσιαστικά ψευδισπόθη και δεν ε, εξυπηρετούν καθόλου το το θεσμικό όργανο που ε, υπηρετούμε. Και πολύ συχνά ε, υποβάλλονται τόσο ακραίες προτάσεις ε, ή κανείς επικεντρώνεται και μεγεθύνει συγκεκριμένες παραγράφους και ουσιαστικά απορρίπτει το σύνολο της έκθεσης. Σίγουρα ε, είναι σημαντικό να εκφράζουμε επιθυμίες και φιλοδοξίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεπερνάμε τις αρμοδιότητές μας. Επίσης, ε, ε μερικοί αναφέρθηκαν στο σεβασμό της Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Α, δεν ε, τίθεται καν αυτό το ζήτημα. Ο χάρτης του το ΟΗΕ γίνεται σεβασμός και γίνεται σεβαστός και η πολιτική ασφάλεια και άμυνα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτει στο χάρτη. Καμία στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωση δεν, νοεί, δεν νοείται χωρίς σεβασμό του χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν τίθεται καν ζήτημα. Δεν χρειάζεται να συζητάμε το θέμα αυτό. Είναι αυτονόητο ότι σεβόμαστε το χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το έργο μας ε, ε, περιχαρακώνεται από αυτές τις επιταγές του Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, ε, με καθησυχάζει το γεγονός ότι με κατηγορούν είτε για υπερβολικό υπέρμοχο του ΝΑΤΟ είτε για διάπειρο πολέμιο του ΝΑΤΟ ταυτόχρονα. Η πραγματικότητα είναι απλούστατη σήμερα. 22 από τι 28 χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και μέλη των ΝΑΤΟ και στις συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούμε για την ανάγκη ανάπτυξη αμυντική πολιτική που δεν θα πρέπει να αποκλεί όμω ή να αντιβαίνει στι δεσμεύσει των χωρών σε ό,τι αφορά τη συλλογική άμυνα. Και δεν υπάρχει κάποιο μηχανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι πιο αποτελεσματικό από τον ΝΑΤΟ για την εξασφάλιση τη συλλογική μα άμυνα. Και αυτό είναι σαφέ και ισχύει. Βέβαια δεν μας ικανοποιεί αυτή η κατάσταση στις, ως προς τις άλλες απειλές ασφάλειας. Στην Αφρική, νοτίως της Επίρους μας, και εκεί δεν πρόκειται το ΝΑΤΟ να δράσει. Οπότε η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί, συλλογικά, αλλά και μεμονωμένα από κάποια κράτη-μέλη, είναι να βρεθεί ένα είδο συμπληρωματικότητα. Οπότε να κάνετε δίκη προθέσεων για το γεγονό ότι είμαι υπέρ μια ευρωπαϊκή άμυνα που θα είναι ο ραγό του ΝΑΤΟ δεν έχει νόημα αυτό που λέτε. Είναι τελείως αναδαφικό. Αλλά και το να πούμε ότι ο μόνος ορίζοντας στο μέλλον είναι το ΝΑΤΟ, ούτε και αυτό ισχύει. Θα πρέπει να ξεφύγουμε λοιπόν από, δογματικές, ε, από δογματικά κολλήματα και ιδεολήψεις και να είμαστε πιο ρεαλιστές. Σε ό,τι αφορά την ε, άρθρωση και το συνδυασμό στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αποστολών, σίγουρα η χρειά της έκθεσης μπορεί να είναι υπερβολικά στρατιωτική ή να στρέφεται υπερβολικά στα στρατιωτικά ζητήματα για μερικού. αλλά ουσιαστικά μη στρατιωτικέ είναι οι αποστολές μας. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και σίγουρα δεν είναι ο αδύναμος ε, ο φτωχό συγγενή, οι μη στρατιωτικέ αποστολέ τη ε, ΚΕΠΑ, ε, οι 4.000 ε, μέλη του προσωπικού που ασχολούνται με τα θέματα των αποστολών είναι κυρίω σε μη στρατιωτικέ αποστολέ. Οπότε δεν είναι ο δύναμο κρίκο τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα οι πολιτικέ μη στρατιωτικέ αποστολές. Το αντίθετο. Και τέλο. Λυπάμαι που έφυγε στο μεταξύ ο κύριο Ριβιέρα, θα το ξανασυζητήσουμε. Αυτή η δίκη προθέσεων για την κοινοτικοποίηση τη αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη. Λίγη σοβαρότητα, παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι. 13 δισεκατομμύρια θα δοθούν στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Άμυνα σε μία αιτία. Δηλαδή, λίγο λιγότερο από 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αυτό το θεωρείτε εσεί ε, κοινοτικοποίηση τη Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. αυτό είναι ένα ελάχιστο συμπλήρωμα για να συμπληρώσουμε τις τεχνολογίες που δεν έχουμε, να καλύψουμε το χάσμα των ικανοτήτων μας και να γίνουμε λιγότερο εξαρτημένοι. Γιατί ο κύριος Ριβιέρ θα ήθελε να γίνουμε ακόμη πιο εξαρτημένοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι ήδη είμαστε. Αλλά ουσιαστικά ένα μικρό σμπρόξιμο δίνουμε, μια μικρή όθηση. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υπαγάγουμε την αμυντική μα πολιτική στον έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την κοινοτικοποιήσουμε. Το αντίθετο. Σα ευχαριστώ. Ε, θυμίζω ότι πριν από την, μέχρι την Παρασκευή μάλλον 12 το μεσημέρι πρέπει να υποβληθούν οι τροπολογίες. 25 και 28 Νοεμβρίου στην ΑΦΕΤ και 4 Δεκεμβρίου η ψήφος για να πάει στην Ολομέλεια το θέμα τον Ιανουάριο. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και σας ξαναδίδω την Προεδρία. Παρακαλώ.